Okay, colleagues, good afternoon and welcome. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ένα θέμα έχουμε μόνο στην ημερήσια διάταξη, την οποία όμω πρέπει να εγκρίνουμε. Την έχετε λάβει, έχει δυναμηθεί. Συμφωνούμε με την ημερήσια διάταξη και σας ευχαριστώ. Στο δεύτερο θέμα και μοναδικό τη ημερήσια διάταξη, πολύ σημαντικό όμω. Έχουμε το μέλλον τη Συμφωνία Σκοτωνού και ο τίτλος της συζήτησης είναι προς μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020 έχουμε τον Επίτροπο Μεμίτσα σήμερα ε, και ένα έγγραφο το οποίο από κοινού ε, μεταξύ Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου δημοσιεύτηκε. ίσως για τους πιο καινούριους να σας, τον σκοπό να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το ιστορικό. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση μεταξύ κρατών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρική Καραϊβική ε, Ειρηνικού, ανάγεται στο, στην πρώτη συμφωνία του 1975. Ακολούθησαν αρκετέ συμβάσει ΛΟΜΕ και στη συνέχεια μια νέα συμφωνία εταιρική σχέση, η οποία εκπνέει το 2020. Η Συμφωνία Κοτονού έχει σε κύριου στόχου, τη μείωση τη φτώχεια, την εφόρο ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των κρατών και στην παγκόσμια οικονομία σταδιακά. Για να βρείτε το πλαίσιο που περιλαμβάνει το εμπόριο, την οικονομική συνεργασία και πολιτικό διάλογο, δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της, ε, το κράτος δικαίου, την χρηστή διακυβέρνηση. Και έτσι Έχουμε ενισχύει τη Συμφωνία Κοτονού εδώ και 15 χρόνια, εκπνέει σε 5 χρόνια και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία όπου συζητούμε εάν τη διατηρούμε, εάν την αντικαθιστούμε, εάν είναι ακόμη επίκαιρη και πρέπει να διατηρηθεί. Με χαρά λοιπόν καλώς ορίζω εδώ τον Επιτροπό Μιμίτσα για να μας παρουσιάσει ένα άγραφο διαβουλεύσεων που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε πολύ ο κόσμος, Επίτροπε από την υπογραφή της τελευταίας συμφωνίας. Έχουν αλλάξει και εμπορικέ σχέσεις. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για παγκόσμιες εμπορικέ σχέσεις, τώρα περνάμε σε περιφερειακές, επί του νέα θεματολόγιο για την ανάπτυξη που συμφωνήθηκε στη Νέα Υόρκη πριν από τρεις εβδομάδες και έτσι θα ήθελα εσείς να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο μέλλον και πώς εγγράφεται σε αυτό το μέλλον της Αναπτυξιακής Πολιτικής Συμφωνία του Κοτονού. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο και μετά θα ακούσουμε και τους βουλευτές για ερωτήσεις και σχόλια. Παρακαλώ. Βεβαίως έπρεπε να καλωσορίσω, όφιλα να καλωσορίσω και τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Συνεργασίας για την Ανάπτυξη, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι παρόν εδώ. Ο κύριος Μιμίτσα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βουλευτές, με χαρά σας βλέπω εδώ για να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για ένα από τα μεγάλα στρατηγικά θέματα που θα μας απασχολήσουν στα επόμενα χρόνια. που σημαίνει να δώσουμε απαντήσει στον τρόπο με τον οποίο θα αναδιαμορφωθούν οι σχέσει μα με τι 79 ε, χώρε Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικού. Η συμφωνία του Κοτονού είναι μοναδική γιατί προσφέρει βάση για συμβατικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 79 αυτών κρατών που ε, αναπτύσσονται σε τρεις διαφορετικές υπήρους. Είναι μια εταιρική σχέση, συμφωνία εταιρική σχέσης και ως εκ τούτου η αναθεώρησή της ε, εγείρει κρίσιμα και στρατηγικά ζητήματα. Έχει να κάνει δηλαδή με τον ρόλο της Ευρώπης στο στο παγκόσμιο σκηνικό, με μεγάλο μέρος των κρατών και πέραν των στόχων της ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε διαρωτώμενοι ποιοι είναι οι στόχοι και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Ιφίλιο και βέβαια έναντι των κρατών αυτών ειδικότερα και πώς μια εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή αυτών των ε, φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δραματίσει ρόλο πρωταγωνιστικό στο παγκόσμιο σκηνικό με έμφαση στις εμπορικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, στις 6 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πατή Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Ασφάλεια, Πολιτική Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν ένα έγγραφο, κοινό έγγραφο διαβουλεύσεων για τις εταιρικές σχέσεις και το μέλλον τους ε, εταιρικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ανοιχτή προς ιονδήποτε ιδιώτη ή φορέα μέχρι το τέλος του έτους. Το έγγραφο καλύπτει πάρα πολλά θέματα, εκφράζει πολλές προσδο... εκφράζονται πολλές προσδοκίες από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και η Επιτροπή με απόλυτη διαφάνεια θα επεξεργαστεί και θα εργαστεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να περιγράψουμε το φάσμα, ως το δυνατόν ευρύτερο φάσμα των ζητημάτων, 23 εν όλο ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από αυτό το έγγραφο των διαβουλεύσεων, με διτούς στόχους που αντιστοιχούν και στα δύο επόμενα βήματα που σκοπεύει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας εκθέσω αργότερα. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να συλλέξουμε στο δυνατόν ευρεία και ει βάθο αξιολόγηση και εμπειρία από τα 15 χρόνια της εταιρική σχέση Κοτονού. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία τη, με την ικανοποίηση των στόχων τη, εάν αυτό δεν επετεύχθη γιατί, Έχουμε ερωτηματικά σχετικά με το πόσο ήμασταν υπερβολικά φιλόδοξοι ή, μήπως, ή εάν υπάρχουν κάποιοι τομεί στου οποίου είχαμε καλύτερε επιδόσει, ενώ κάποια, σε κάποιου άλλου είχαμε χειρότερε. Πόσο καλά λειτουργήσαν οι μηχανισμοί τη συμφωνία. Και δεύτερον, αναζητούμε ιδέε, προτάσει, σχόλια από του εταίρου για να οικοδομήσουμε μια στρατηγική προ το μέλλον. Ω εκ τούτου, έχουμε Ω ερώτημα για το μέλλον, πώ μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον, σε ποια ζητήματα πρέπει να εστιαστεί με μελλοντική εταιρική σχέση, αν πρέπει να ανοίξει συμφωνία και προ άλλε χώρε, αν πρέπει να περιοριστεί σε ορισμένε μόνο χώρε, εάν ε, θέλουμε να εισαγάγουμε και, την, ε, και το καθεστώς του παρατηρητή, εάν ε, η ΑΚΕ είναι ο καλύτερο εταίρος δεδομένου ότι έχει αλλάξει πολύ ο, κόσμο κόσμος τα τελευταία 15 χρόνια, ή αν πρέπει να παραμείνει ως δεσμευτικό εργαλείο, ή αν υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ. Στα περισσότερα από αυτά ερωτήματα και αυτά που κοιτάνε προς το παρελθόν και αυτά που στρέφονται προς το μέλλον, προσπαθούμε να καταγράψουμε δεδομένα για το περιεχόμενο και την ε, δομή τη εταιρική σχέση. και προσπαθούμε να συλλέξουμε συνεισφορέ από πολυάριθμες και διαφορετικέ πηγέ και βέβαια θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για να αξιολογήσουμε την κάθε πρόταση τη επιμέλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Σχέσης παράλληλα αναπτύσσουν και εσωτερικό διάλογο. Οι επικεφαλεί των ε, αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κράτη ΑΚΕ, θα αναπτύξουν διάλογο για το παρελθόν και δεχόμενο μέλλον της εταιρικής σχέσης και σε εθνικό επίπεδο και θα καλέσουν όλους τους εμπλεκόμενους στην κάθε χώρα φορεί. και βεβαίως αυτά όλα θα ενσωματωθούν στην αναλυσή μας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στο στάδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική δράση δεν έχουν προεπιλέξει αδίποτε λύση. Ε, παραμένουμε ανοιχτοί σε όλε τι προτάσεις, δεν έχουμε ακόμη ε, αποφασίσει ως προς τις προτάσεις που θα διατυπώσουμε και θα υποστηρίξουμε. Αυτή η διαβούλευση είναι και η καλύτερη δυνατότητα που έχουμε για να αναπτύξουμε τις ιδέες μας. Ωστόσο υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Η εταιρική μας σχέση με τις χώρες ΑΚΕ ξεπερνάει τα τελευταία 15, 15 ετία. Έχουμε ξεκινήσει από το 1975 τις ε, συμφωνίες, ωστόσο οι σχέσεις μας με τα κράτη-μέλη, με τα κράτη ΑΚΕ, ε, ανάγονται στις απαρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 60 χρόνια πριν δηλαδή. Τα κράτη ΑΚΕ και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το όλων 110 χώρες, έχουν και την πλειονοψηφία στα Ηνωμένα Έθνη. Η εταιρική αυτή σχέση αποτελεί και τη δύναμη αλλά και την ευκαιρία, ε, μια μεγάλη ευκαιρία που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε η Συμφωνία Κοτονού είναι μοναδική ω προ την ουσία τη. αντίστοιχη δεν υπάρχει διεθνή συνθήκη δηλαδή που να μπορεί να συγκριθεί μαζί τη. Έχει περιεχόμενο πολύ φιλόδοξο, ε, αναπτύσσει μια σειρά αποζητημάτων που πάνω απ' όλα έχουν σαν στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας στις πιο φτωχέ χώρες του κόσμου. Οι χώρες που πριν από 15 χρόνια συνήθισαν τη συμφωνία έχουν αλλάξει ουσιοδός έκτοτε. Αφενός μεν έχει διπλασιαστεί ο αριθμό των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτεραιότητες των νέων κρατών μελών θεμητά δεν είναι οι ίδιες όπως πριν από 15 χρόνια. Από την άλλη κάθε κράτος ΑΚΕ έχει εξελιχθεί κατά διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο και αυτό πρέπει να αξιολογηθεί με ακρίβεια. Και τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των κρατών αυτών έχουν αλλάξει στον χρόνο. Συγκρινώντα λοιπόν αυτά τα συμφέροντα, δεν πρέπει να λησμονούμε ένα πολύ απλό γεγονός ότι μερικά από τα κράτη-μέλη μας έχουν εισόδημα κατά κεφαλήν χαμηλότερο από ορισμένα από τα κράτη ΑΚΕ. Ως προς το πεδίο εφαρμογή της συνθήκης, συμφωνίας, κάποια από τα ζητήματα προτεραιότητας έχουν αντιμετωπιστεί, κάποια παραμένουν, κάποια είναι ακόμη πιο προβληματικά και ανησυχητικά και έχουν προσθεθεί και νέα ζητήματα η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η μετανάστευση, η ειρήνη και η σταθερότητα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εξάπαντος πρέπει να αποτελέσουν τμήμα των κοινών προτεραιοτήτων μας. Επιπλέον αυτού, η σημασία των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων συγκρινόμενη με την αναπτυξιακή βοήθεια είναι πολύ σημαντικός παράγον και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε παράλληλα. Η αρχή τη επικουρικότητα ασφαλώ θα δραματίσει σημαντικό ρόλο σε ορισμένε πτυχέ και στι πτυχέ αυτέ πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί με μία φωνή. Πέραν τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών ΑΚΕ, παράγοντε στον χώρο του εμπορίου και της ανάπτυξης ε, είναι διαφορετικοί. Έχουμε οικονομίες ε, οι οποίε διαδραματίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο σε διαφορού τομεί, αναπτύσσονται διαφορετικά συμφέροντα και εταιρικέ σχέσει. Πρέπει να καταγράψουμε λοιπόν την ε, νέα αυτή κατάσταση και να αναλογιστούμε ποιες είναι οι τάσεις που μπορεί να ακολουθήσουν τα κράτη και οι περιφέρειες τι επόμενες δεκαετίες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το μελλοντικό πλαίσιο ενισχύει και δεν αποδυναμώνει τις σχέσεις μας και το ρόλο μας. Η βιώσιμη φόρη ανάπτυξης και ε, το θεματολόγιο για την ανάπτυξη καθορίζουν ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα πρέπει να προσδιοριστεί και η αναπτυξιακή μας πολιτική, αλλά και όλες οι διεθνείς μας δεσμεύσεις. Πρέπει να παρακολουθήσουμε, να συζητήσουμε με βάση αυτές τις αρχές. Η ευελιξία των εργαλείων που θα αναπτύξουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης η υπογραφή της Συμφωνίας Κοτονού αλλά και η κύρωση των τροποποιήσεων της αρκετά χρόνια και αυτό οδήγησε σε δυσκολίε. Πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει. Σε ευρύτερη έννοια, θα ήθελα να καταστήσω ένα σημαντικό ζήτημα, ότι αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να επισημάνει και τις ε, αδυναμίες του τρόπου εργασίας μας. Δεν θα διστάσω να προβώ και σε αυτοκριτική. Ε, αναφέρομαι βέβαια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κοινά όργανα αλλά και τους μηχανισμούς που έχουμε αναπτύξει στην εργασία με τους εταίρους μας. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε πώς οι ίδιοι εταίροι έχουν εργαστεί, τι είδους επιδόσεις είχαν και πόσο τήρησαν τους κοινούς στόχους ή υλοποίησαν τους κοινούς στόχους. Συμπεράσματα και διδάγματα για το μέλλον θα πρέπει να διατυπωθούν και βέβαια για το κοινό στόχο που θα πρέπει να επιδιώξουμε με στόχο την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τα μελλοντικά βήματα τώρα. Αυτό το κοινό έγγραφο διαβουλεύσεων είναι το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό έγγραφο για σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης. Περαιτέρω βήματα όμως, ε, αλλά και ε, επαφές και επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναπτυχθούν ε, στο επόμενο έτος, στο δε πρώτο τρίμηνο του 2016 και επί τη βάση αυτής της δημόσιας διαβούλευσης και του ιστορικού διαλόγου θα καταθέσουμε μια πρώτη αξιολόγηση, άτυπη αξιολόγηση της πρώτης 15 ετίας ε, ισχύως της Συμφωνίας Κοτονού, στην οποία θα εκτίθενται οι κύριοι πυλώνες της Συμφωνίας με βάση αποδεικτικά και στοιχεία για να διατυπωθούν συμπεράσματα από αξιόπιστες ε, πηγές και δεδομένα. Σε δεύτερο επίπεδο θα γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου με καταγραφή όλων των επιλογών που μας απασχολούν και πάλι βάση των διαβουλεύσεων στόχος θα είναι η περιγραφή και αξιολόγηση διαφορετικών ενδεχομένων και σενάριων και των πιθανών συνεπειών τους. Πέραν αυτού και περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΠΑΤΗ εκπρόσωπος θα καταρτήσουν μια κοινή ανακοίνωση όπου θα περιγράφουν αναλυτικά τη στρατηγική που σκοπεύουν να αναπτύξουν. Ε, όπως βλέπετε υπάρχουν διαφορετικές και αρκετές δυνατότητες για συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βέβαια και εγώ θέλω να συνεργαστούμε στενά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλώς εκ παραλλήλου θα ε, διαβουλευτούν με τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο, τα κράτη και έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι είναι συγκλίνοντα τα συμφέροντα και βεβαίως θα έρχομαι να σας ομιλώ όποτε θεωρείτε σκόπιμο για το θέμα αυτό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω να ακούσω και τις δικές σας αντιδράσεις. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρουν οι ε, επόψεις σε σχέση με το ποιε θεωρείτε τις μεγαλ... ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την ε, νέα αυτή προσπάθεια. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι στόχος μας είναι να γίνει η Φίλες ένας καλύτερος τόπος όπου θα ζούμε όλοι μαζί και ιδιαίτερα θα είναι καλύτερος τόπος για αυτούς που φέρουν το πιο πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ευχαριστούμε που από την αρχή της διαδικασίας κοντά μας για να ξεκινήσουμε αμέσως στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται πολύ ε, σκέψη για να δούμε τι μορφή θα πάρει αυτή η μελλοντική εταιρική σχέση. Έχουμε εντοπίσει αυτό το θέμα ως μια από τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας για την ερχόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια βέβαια. Έτσι όπως περιγράψετε άλλωστε τη διαδικασία η πρώτη φάση των διαβουλεύσεων είναι σύντομη, έξι εβδομάδες, 8 ε, μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αντιδράσει σύντομα και βεβαίως θα το συζητήσουμε σε επίπεδο συντονιστών, αλλά πρωτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ξέρουμε πότε θα ε, δημοσιευτεί ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Yeah, so anyway, we, we, we can, we Εντάξει λοιπόν, οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο. Θα έχουμε την ε, αξιολόγηση με τη μελέτη εντεκτύπου. Θα υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία να τα αναμένουμε. Ωραία, όταν ξαναέρθετε θα μας εξηγήσετε τι θα γίνει με τη μελέτη αντικτύπου ή τις υπόλοιπες επιλογές. Η ανακοίνωση φαντάζομαι ότι θα παρουσιάζει την απόφαση, του στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα υπάρχουν κάποιε επιλογέ και μετά εθνικέ προτάσει. Έτσι σκοπεύετε να προχωρήσετε, μάλλον. Ο κύριος Τιε για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσίαση τις διαδικασίες διαβουλεύσεων και για το έγγραφο. Είναι πραγματικά πολύ ανοιχτό μια προσέγγιση και πολύ έντιμη με την παρουσίαση των διαφορών επιλογών και εντοπίζει τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν και στο μέλλον σε σχέση με τη Συμφωνία Κοτονού. Νομίζω το θεματολόγιο του 2030 είναι το προφανές πλαίσιο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συζητούμε το μέλλον της Συμφωνίας Κοτονού και υπ' αυτήν την έννοια έχουμε πλέον νέους στόχους. Δεν είναι μέρος των στόχων της χιλιετίας, του πλαισίου MDG, αλλά έχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης 16. Ήδη λοιπόν μέσω του πολιτικού διαλόγου απηχείται εν αυτό στη Συμφωνία Κοτονού. Πρέπει να ενισχυθούν ωστόσο και στο μέλλον. Μιλάμε για ειρήνη και ασφάλεια, καλή διακυβέρνηση, οι διαστάσεις αυτές εντοπίστηκαν και από μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των αιτίων της διαφθοράς και κατά της ανάπτυξης και διαπιστώθηκε ότι στις χώρες ΑΚΕ είναι εξυπηρετούν τα που χρησιμοποιούμε στις δικές μας πολιτικές, στις εθνικές διαδικασίες ή στις πολιτικές γειτονία. Οπότε, δεν λέω να κάνουμε copy-paste αναγκαστικά, αλλά κάποιες από αυτές τις ε, εμπειρίες και τους πειραματισμούς να τα εκμεταλλευτούμε για να ενισχύσουμε την προσέγγιση μας. Είναι λοιπόν ε, πολύ καλή σύμπτωση που ο ίδιος ο Επίτροπος προσωπικά είναι πλάκη στις διαδικασίες αυτέ, γιατί γνωρίζει και τη διαδικασία ένταξη τη Κροατία λόγω χάρη και ξέρει πολύ καλά του συγκριτικού δείκτε για κεφάλαια όπω ε, η δικαιοσύνη, η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Βεβαίω, ο διάλογο για τη μετανάστευση είναι κάτι που είναι επίκαιρο σήμερα, αλλά θα μα απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και την ερχόμενη δεκαετία ολόκληρη. Μιλάμε για, την, για διάλογο σε σχέση με πανεισδοχές, με καταπολέμηση λατρεμπορίας. Είναι και αυτό μία από τις πτυχές που θα θέλαμε να ενισχυθεί στο μέλλον. Μετά οι θεσμικές πτυχές. Δεν έχω σαφή εικόνα ακόμα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Η πιο απλή θα ήταν να διατηρήσουμε το πλαίσιο ακαίο όπως ισχύει με μια αρχή διαφοροποίησης. Δηλαδή με κάποιες ε, εναλλαγές ανάλογα με το αν πρόκειται για τον Αφρική ή τον Ειρηνικό αλλά κάποιες σκληρές ερωτήσεις ε, για το θέμα της πολιτικής βούλησης πρέπει να τις θέσουμε δηλαδή η μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση, η κοινοβουλευτική διάσταση σε όλα αυτά. Ξέρω ότι θα οργανωθεί μια τέτοια σύνοδο τον ε, Δεκέμβριο, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει το μέρο. Είναι θέμα διοργανωτικό μεν, αλλά δείχνει τι επίπεδο πολιτικού ενδιαφέροντα μπορεί να υπάρχει, τι πολιτική βούληση για να οργανωθούμε γέρο. και δεν έχουν οργανώσει οι εναλλασσόμενε προεδρίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μεικτέ κοινοβουλευτικέ συνόδου στα κράτη του εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν να μα απασχολήσει αυτό από θεσμική πλευρά. Και τελευταία παρατήρηση. Μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα την ακούσετε, ούτε και τελευταία, για την αναπτυξιακή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εκτός του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού θα ξέρατε ότι για μας το ιδανικό θα ήταν να βρίσκεται εντός του προπολογισμού, απλώς ήθελα να το επαναλάβω για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και με τους συναδέλφους της Μικρής Κοινοβουλευτικής για το θέμα αυτό. Ο Γκερέρο. Ο Γκερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Μίμητσα και για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή μας και για την ενημέρωση που μας έκανε για αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Έχει δεσμευτεί λοιπόν πλέον ε, η Επιτροπή, ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Μας ενημέρωσε όμως ο Επίτροπος και για τα επόμενα στάδια στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας να δούμε και εμείς ε, ως Κοινοβούλιο και συγκεκριμένη δική μας Επιτροπή πώς μπορεί να παρέμβει σε καθένα από αυτά τα στάδια. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια. Καταρχάς, Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που θεωρούν ακόμη ότι είμαστε πολύ μακριά από την αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού. Τέσσερα και χρόνια Ίσως μάλιστα να υπάρχουν και κάποιοι ε, βουλευτές ε, που θα πιστεύουν ότι δεν θα είναι πια βουλευτές όταν γίνει αυτή η αναθεώρηση. Και έχουν χάσει κάπως το ενδιαφέρον τους για την όλη διαδικασία. Πάντως αυτό το οποίο μας διδάσκουν όλες αυτές οι σύνοδοι κορυφής ε, που βλέπουμε αυτή τη χρονιά σε σχέση με τους στόχους, ε, τους αναπτυξιακούς κτλ. δείχνουν ότι οι αλλαγές, ε, οι σύνοδοι κορυφής, οι αναθεωρήσεις ε, χρειάζονται χρόνο προετοιμασίας. Αυτό πρέπει να γίνει εκ των προτέρων. Άρα σωστό είναι να έχουμε υπόψη μας το 2020 ως χρονικό ορίζοντα. Και επίσης είναι πολύ σωστό που ακολουθήθηκε αυτή η επιλογή της διαδικασίας διαβούλευσης όλες οι μεγάλες συνεδριάσεις που έγιναν φέτος έχουν κάποια προηγούμενα, διαβουλεύσεις δηλαδή. Ε, και η Σύνοδος Κορυφής για τα ανθρωπιστικά ζητήματα που θα λάβει χώρα του χρόνου είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτατης διαδικασίας διαβούλευσης. Ολοκληρώθηκε στη Γενέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η γενική διαβούλευση και νομίζω ότι μεγάλες αλλαγές που έχουν επισυμβεί και επισυμβαίνουν στις κοινωνίες μετά την έγκριση πρώτης συμφωνίας Κοτονού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την ανάδυση μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, μιας ισχυρής δομής οργανώσεων αναπτυξιακής συνεργασίας, συνηγόρων, μάλλον υπερμάχων των δικαιωμάτων, ανθρώπων που είναι υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης κτλ. κτλ. Και αυτό σίγουρα υπερβαίνει τις απλές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών ή τις διαπεριφερειακές συμφωνίες διαφόρων μορφών. Άρα, καλό είναι που υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Τώρα θα στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, όπως θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε αυτό το πλαίσιο ή σε πλαίσιο των κρατών μελών, όπως είπε ο Επίτροπος ε, Μίμητσα, καλό θα ήταν. Και ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διοργάνωσης ε, κοινή διαβούλευσης, δηλαδή μεταξύ χωρών ή οργανώσεων ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν ένα τμήμα της αξιολόγησης του πώς ε, λειτουργήσε η συμφωνία τα τελευταία 15 χρόνια και ποιες είναι οι προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωπες και ποιες είναι οι επιθυμίες μας για το μέλλον. Καλό θα ήταν αυτά όλα να μην γίνουν χωριστά από, τους, τις δύο πλευρές, από τη μία Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη χώρες ΑΚΕ, αλλά καλό θα ήταν πιστεύω σε κάποια χρονική στιγμή να έχουμε κάποιες γέφυρες και κάποια κοινά σημεία για να μπορέσουμε να εξολογήσουμε από κοινού την κατάσταση. Σε αυτό του λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο και το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Και θα είναι ακόμα πιο σημαντικό μέχρι το 2020. Δηλαδή, η Συμφωνία ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποια θέση θα τοποθετηθεί, αν θέλετε, στο ε, πλαίσιο όλων αυτών των συμφωνιών που ε, συζητούνται. Έχουμε την εμπορική συμφωνία με τον Ειρηνικό που βρίσκεται στη φάση της επικύρωσης αυτή τη στιγμή. Αν προχωρήσουμε έχουμε και άλλες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, έχουμε το TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν όλες αυτές οι συμφωνίες πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών. Ιδίω για χώρε που θα μπορούσαν να είναι συμβαλόμενα μέρη ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιφερειακέ συμφωνίες. Θα μπορούσαν, παραδείγματο χάρη, κάποιε χώρε να υπογράφουν ε, την ε, συμφωνία για τον ειρηνικό, αλλά και τη συμφωνία Κοτονού. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τα κοινά σημεία και να αποφύγουμε αντιπαραθέσεις η εμπειρία μου ως μέλος ε, της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Εκπροσώπησης μου διδάσκει ότι το πιο προβληματικό αν θέλετε στοιχείο αυτών ε, που κάναμε τα τελευταία 15 χρόνια ήταν οι εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες. ΕΠΑ. Δηλαδή συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Κλασικό. Στις συνεδρίες Ευρωπαϊκή Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει λοιπόν στις εργασίες μας, να το σκεφτούμε και να επαναπροσδιορίσουμε το σημείο αφετηρίας μας. Όλα αυτά σχετίζονται και με τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που αυτή τη στιγμή, ε, σε αυτή την ιστορική περίοδο, ε, έρχονται προς το μέρος μας. Δεν θα πάψουν και δεν θα μειωθούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το πρόβλημα στη ρίζα του. Και αυτή θα είναι για μας η μεγάλη πρόκληση και από την άποψη της δουλειάς μας και τη συνεργασία μας με τις χώρες ΑΚΕ στην περίοδο μετά το 2020 και στις συζητήσεις που ήδη έχουμε κάνει στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση για ένα θέμα που είναι προσφυλές για μένα. Τις ε, περιφέρειες για τα διαμερίσματα τα υπερπόντια. Ξέρετε ότι αυτές οι περιφέρειες έχουν το δικό του νομικό καθεστώς ως το 2020. Στην απόφαση σύνδεσης των ε, περιφερειών των υπερποντίων είναι μια απόφαση του 2014. Η ερώτηση μου είναι, εάν σκοπεύετε να προτείνετε κάποιο ιδιαίτερο δημοσιονομικό εργαλείο για τις ε, περιοχές και τα διαμερίσματα που είναι εξωχώς απομακρυσμένα, τις υπερπόντιες δηλαδή αυτές ζώνες. Πρόκειται να προτείνετε κάποιο ειδικό εργαλείο για τις χώρες αυτές, τις υπερπόντιες περιφέρειες και διαμερίσματα. είναι μέρο τη κοινωτική επικράτεια. Αλλά αυτό το εργαλείο θα το υποβάλλετε και στο Κοινοβούλιο και στου βουλευτέ για να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε κυρία Ρενά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καταρχάς ευχαριστούμε για τη διαδικασία διαβουλεύσεων που προτείνατε. Είναι σημαντικό να διευρύνουμε να ακούσουμε, να φουγκραστούμε τα όσα συμβαίνουν από την πλευρά των Αφρικανών εταίρων. Είναι σημαντική διαδικασία και σας ευχαριστούμε για αυτή. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε με τη Γενική Διεύθυνση Τρέντ για το θέμα των ε, χωρών ΑΚΕ και τις οικονομικές, τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να το συζητούμε και εδώ. Όπως θα ξέρετε, οι πολυμερείς διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΠΟΕ έχουν πάψει, διότι χώρες του Νότου δεν μπορούσαν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε αυτές τις ε, μεγάλες εμβέλειες οικονομικές ε, πολυμερείς συμφωνίες. Η απόκριση σε αυτήν την ε, πάυση σε επίπεδο ΠΟΕ είναι οι διμερείς συμφωνίες, που όμως δεν λαμβάνουν αναγκαστικά υπόψη τις μέρημνες των χωρών του Νότου. Ξέρετε ότι τώρα διαπραγματευόμαστε την Διατλαντική ε, Συμφωνία που θα έχει επιπτώσει και στην Αφρική, όμω σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψει των Αφρικανικών χωρών. Δεν σκεφτόμαστε τι μπορεί να συμβεί τι Αφρικανικέ χώρε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών μα για τον πίκτη. Έτσι λοιπόν ελπίζω η Επιτροπή από τη δική σα την πλευρά κύριε Μελθέ να μπορέσει να χάρη τη δική σα παρέμβαση να ευαισθητοποιήσει όλου του Επιτρόπου, του Επιτρόπου οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο για να υπάρξει συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή αυτά που δίνουν σε αφρικανικέ χώρε από τη μία να μην από την άλλη ε, με τι διεθνεί μα συμφωνίε. Τώρα για τι χώρε μιλάμε για αλληλεγγύη για αμοιβαιότητα με τις χώρες ε, ΑΚΕ. Βλέπουμε ότι όταν μιλάμε για χώρες, τις πλέον χώρες στον κόσμο, 26 από αυτές είναι χώρες που έχουμε τέτοιες συμφωνίες από τις οποίες ζητούμε αμοιβαιότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι από, αναπτυξιακής, από αναπτυξιακής πλευράς είναι στη επίπεδο με εμάς. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις διαφορές στην οικονομική μας προσέγγιση με τις χώρες αυτές ω προ τι χώρε αυτέ μάλλον. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι σχέση είχατε ω υπέρμαχος της ανάπτυξης ε, σε σχέση με τους συναδέλφου σας, ιδίω αυτούς που ε, ασχολούνται με τα εμπορικά θέματα και πώς καταφέρατε να τα εξισορροπήσετε κάνοντας, ε, βρίσκοντας την σωστή αναλογία και χωρί να πλήττονται οι μένει βάρο των δε. Και για τις περιφερειακές διαιρέσεις και διχασμούς που υπάρχουν. Ενώ η Συμφωνία Κοτονού προέβλεπε την ε, περιφερειακή ολοκλήρωση και ένταξη, πώς θα μπορούσαμε αυτό να το επιδιώξουμε περισσότερο, χωρίς να υπάρχει και άλλη διαίρεση όπως προβλέπουν οι, οικονομικές, οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής Και τέλος, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα παράδειγμα, το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει καμία αναφορά, καμία μνήμα. Αυτό καλύπτεται ελάχιστα στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Δεν θα μπορούσατε να αναλάβετε λοιπόν εσείς αυτό το λάβαρο, να το σηκώσετε και να πείτε ότι σε κάθε περίπτωση συμφωνιών πρέπει και το, η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καλύπτεται. Και πάλι για να επαναλάβω στο θέμα της αμοιβαιότητας, την περασμένη εβδομάδα με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου μας έλεγαν θα υπάρξει ε, αναστολή των τελειωνικών δασμών, ε, δηλαδή κατάργησή τους. Στον προπολογισμό των Αφρικανικών χωρών όμω, αυτή η τελωνική δασμή είναι ένα σημαντικό έσοδο που τους επιτρέπει να επενδύσουν σε κρατικές πολιτικές τους. Κάποιοι θα πούνε, ναι, αλλά στα τελωνία υπάρχει πολλή διαφθορά. Εντάξει, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα και σίγουρα θα πρέπει να επιληθεί το θέμα τη διαφθοράς. Αλλά αν υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους από ένα υπολοιπόμενο κέρδο από τους κρατικούς προπολογισμούς, θα πρέπει να το σκεφτούμε πώς θα ε, αντισταθμιστεί αυτό. Οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου μας έλεγαν μην ανησυχείτε, δεν θα προβλέψουμε εμείς την αποζημίωση για την κατάργηση των πετρελαϊκών δεσμών, θα γίνει αυτομάτως από την λειτουργία της αγοράς. Ε, κάποιοι πιστεύουν ότι η αγορά μπορεί να τα λύσει όλα μόνη της. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, δεν ανήκω σε αυτούς. Ε, σε κάθε περίπτωση αν κάτι επιλύσει αυτό μπορεί να γίνει πολύ μακροπρόθεσμα. Ίσως λοιπόν αργότερα να υπάρξουν διορθώσεις μέσω της αγοράς που θα μειώσουν τις τιμές κάποιων τροφίμων για του Αφρικανού, αλλά δεν νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα θα επιληθεί έτσι το πρόβλημα. Θα ήταν λοιπόν καλό να υπάρχει μια διαδικασία αντιστάθμιση, ε, αποζημίωση, που κάτι θα δώσει σε αυτά τα αφρικανικά κράτη που θα χάσουν από την κρατικά του έσοδα. Και άλλη μια παρατήρηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σαφέ ότι η Συμφωνία Κοτονού μιλάει πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα αναρωτηθεί κανεί. Μήπω πρέπει να ξαναδούμε το άρθρο 96 την ε, περίπτωση παραβιάσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων από τις χώρες, τις συμβαλόμενες Όμω, το είπε και ο Ιταλό συνάδελφο αμέσω πριν, θα πρέπει να δούμε και τα θέματα διακυβέρνηση, όχι μόνο από τη σκοπιά ε, των κυβερνήσεων. Φυσικά είναι ευθύνη μια κυβέρνηση η καλή διακυβέρνηση μια χώρα. Είναι όμω και η διακυβέρνηση των πολυεθνικών να έχουν την σωστή διακυβέρνηση. Όταν κάποιε πολυεθνικέ εκμεταλλεύονται φυσικού πόρου σε χώρε όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοιχνεύσει κανεί ακριβώ το τι εκμεταλλεύτηκαν στη συγκεκριμένη χώρα, ε, η καλή διακυβέρνηση πρέπει να στηρίζεται και στη δική του ε, συμπεριφορά και διαγωγή. Πώ λοιπόν στα πλαίσια τη Συμφωνία Κοτονού μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ανάληψη ευθύνη από τι πολυεθνικέ, διότι ξέρουμε ότι από την άποψη του ε, ΑΕΠ οι πιο φτωχέ χώρε είναι συνήθω αυτέ που έχουν του περισσότερου φυσικού πόρου. Πρέπει και αυτό να επιχειρήσουμε να το επιλύσουμε μέσω των συμφωνιών κοτονού. Και θα πρέπει κάπως μια διάσταση ανθρωπιάς να προσθεθεί και στις εμπορικές μας προτεραιότητες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος... Σάρλ Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τις τέως βρετανικές, γαλλικές, γερμανικές, πορτογαλικές απικίες κυρίως μεταξύ των χωρών και ε, κυρίως έτσι. Και τελικά το σύνολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνει ένα είδος ε, κοινοπολιτείας. Είναι σαν να είναι ένα Commonwealth Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε με αυτό το προνομιακό πλαίσιο σχέσεων θετική εμπειρία δεν υπήρχε, έπρεπε να το εφεύρουμε. Δύο δυνατότητε έχουμε τώρα. Ή θα διαπραγματευτούμε μέχρι το 2020 μια νέα συμφωνία, ή δεν θα τα καταφέρουμε να έχουμε διαπραγματευτεί μια συμφωνία μέχρι το 2020. Την πρώτη υπόθεση, δηλαδή μη συμφωνία, τι θα γίνει πριν τα τέλη του 2019 θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ένα μικρό πρωτόκολλο για να δούμε τι θα γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, γιατί κάποιοι, ε, κάποιοι πόροι θα έχουν μείνει ε, ανεκμετάλλευτοι μέχρι το τέλος του 19. Από εκεί και πέρα, τα κράτη-μέλη τη Ένωση, ε, έχοντα δεσμευτεί ε, σε σχέση με ένα επίπεδο χρηματοδότησης που μπορεί να είναι της τάξης του 0,5-0,6 γιατί ε, έχουμε αναβάλει το 2030 ε, το 0,7% στόχο χρηματοδότησης. Οι χώρες αυτές δεν θα χρηματοδοτούν πλέον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Και τι θα γίνει τότε. Θα έχουμε πάντοτε, αν από δημοσιομίσεις να δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου κανείς δεν θα θέλει να πάει πάνω από το 1% ε, στο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αν αφαιρέσουμε τα, ταμί, τα κονδύλια του ΕΤΑ, ή τέλο πάντων αν δεν υπάρχει καν Ευρωπαϊκό τέμα Ανάπτυξη, πώ θα εκμετευθούν ε, οι πόροι αυτοί, γιατί μέχρι στιγμής η Κομισιόν είναι αυτή η οποία είναι ένα είδο εκτελεστικού οργανισμού για το ΕΤΑ που αποτελεί διοκτησία των 28 κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θα περνάνε τα χρήματα αυτομάτως από τις Βρυξέλλες και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε τα κονδύλια ή τα μέσα για να ε, χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα τα οποία είχαν ε, δαπανηθεί μέσω του ΕΤΑ στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τα βρούμε αυτά τα χρήματα πια, διότι αν το 1% είναι δεδομένο και δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα, τι θα κάνουμε. Αν διατηρήσουν το επίπεδο χρηματοδότησης ε, οι χώρες ε, της Ένωσης, θα το κάνουν από τον εθνικό του προϋπολογισμό. Υπάρχουν χώρες που ε, προσφέρουν λιγότερα και άλλες που προσφέρουν περισσότερο στο ΕΤΑ, εφόσον πρόκειται για θελοντική συμμετοχή. Άρα θα έχουμε ένα σενάριο επανακρατικοποίηση των εθνικών αντιεξοπολιτικών πολιτικών. Και αυτό θα έχει την εξή συνέπεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει μόνο το ίμιστο χρημάτων που διαθέτει σήμερα για τον προγραμματισμό μέσω του DCI ε, δηλαδή του μέσου αναπτυξιακή συνεργασία ή μέσω του ΕΤΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Άρα, ουσιαστικά θα κάνουμε το αντίθετο από ε, το ευκταίο. Για αρκετά χρόνια προσπαθήσαμε να συντονίσουμε καλύτερα τι ε, Ευρωπαϊκέ με τις εθνικές πολιτικές. Τώρα χάνουμε σχεδόν τα μισά λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μα και τα κράτη-μέλη θα κάνουν το καθένα το δικό του εθνικό προγραμματισμό. Αυτό είναι λοιπόν ένα σενάριο που δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Και από την πλευρά της ε, ε, συνοχής, της ε, συνέπειας των πολιτικών θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Δεύτερον, δεύτερο σενάριο, έχουμε νέα συμφωνία και εκεί πρέπει να εγγράψουμε στον προπολογισμό, να, να προβλέψουμε τις δαπάνες. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα διατηρήσουμε τουλάχιστον ε, το υφιστάμενο επίπεδο εσόδων ε, για την Κομισιόν να μπορέσει να εργαστεί. Αν όχι, θα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα πείσουμε τις αφρικανικές χώρες, χώρες του Ειρηνικού και της Καραϊβικής. Alors, le scénario idéal... Το ιδανικό σενάριο θα ήταν, διαπραγματευόμαστε μια νέα συμφωνία, εγγράφουμε τη συμφωνία στον προπολογισμό, προβλέπουμε τα σχετικά κονδύλια με σαφή δέσμευση από τα κράτη-μέλη ότι θα διατηρήσουν το επίπεδο των εκταμιεύσεών του τουλάχιστον στο επίπεδο που θα έχουν φτάσει το 2020. Αν δεν φτάσουμε σε αυτό, δεν θα έχουμε νέα συμφωνία με τι χώρε ΑΚΕ. Δεν ναι, και χαζί. Ε, τα βλέπουν τα πράγματα, βλέπουν πώ ε, λειτουργούν ε, και οι κανόνε εκταμίευση. Άρα θα πρέπει να δώσουμε ορατότητα προβολή. Δεύτερη σκέψη, δεύτερος προβληματισμός. Ε, τι απάντηση θα δώσουμε στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο Κίνα, Ινδία, ε, χώρες που προσλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, με άλλη αιρεσιμότητα θα πρέπει να δούμε τα θέματα της αιρεσιμότητας για μετά το 2020 και το αυτό θα είναι απλή υπόθεση. Και επειδή έχει αλλάξει το πλαίσιο όπως είπα, ήδη σήμερα έχουμε τουλάχιστον 12 χώρες ε, που ε, είναι οικονομικά αναδυόμενες, θα έχουμε και άλλες ε, στο μέλλον, αλλά θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι ανισότητες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε και τα μέσα και τους τρόπους για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αυξανόμενες ανισότητες που υπονομεύουν τι αφρικανικές κοινωνίες. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το πετύχουμε με, με τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, αν εφαρμοστούν σωστά. Τώρα, σε επίπεδο σχέσεων με τις χώρες ΑΚΕ, υπάρχουν κάποια πολύτιμα και Η Συμφωνία Κοτονού ή οι Συμφωνίες Κοτονού που ελπίζω ότι θα παραμείνουν στο Δημικές με τη μια την άλλη μορφή, περιέχουν κάποιες διατάξεις. Συμφωνώ τον Κοτονού λοιπόν περιέχει διατάξεις που μας ε, ε, ενθαρρύνουν να πούμε στους πολιτικούς μας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όλες οι χώρες ε, μέλη και ουσιαστικά πρέπει να έχουν εμάς ως συνομιλητές τα λοιπά. υπέρμαχος ε, του ε, πολυμερού συστήματος. Ε, εάν θέλουμε λοιπόν να υπερισχύει αυτό το σύστημα, χρειαζόμαστε έναν πολύ ισχυρό εταίρο. Και στην εισαγωγική μου παρατήρηση μίλησα για το είδος αυτής της κοινοπολιτείας, αλλά ευρωπαϊκά, το Commonwealth. Οι πορικές συμφωνίες, εάν δώσουμε νέα πνοή, νέα δυναμική στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά 80 χώρες ΑΚΕ, 30 ευρωπαϊκές. Έχουμε ένα G110 που έχει μεγάλο βάρος και στον πολιτικό διάλογο και μπορεί να τυπώνει ξεκάθαρα τους στόχους ε, στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων σε πολυμερή κλίμακα. Οπότε η Ευρώπη θα μπορούσε και αυτή τότε με όλο της ε, το βάρος, ε, με όλη της τη βαρύτητα να επηρεάσει τις συμφωνίες, ε, μια συμφωνία κοτονού νούμερο 2, πείτε τι όπως θέλετε. Και θα μπορούσε αυτό να είναι ένας αμοχλός, να έχουμε μια πιο ισχυρή θέση, ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο προσκήνιο. Έχουμε κοινέ απόψεις, κοινέ αναλύσεις. Νομίζω θα ήταν κρίμα να διακινδυνεύσουμε, να εγκαταλείψουμε μια πρακτική που έχει ε, αποδείξει ότι δουλεύει. Και ε, μπορούμε να μιλάμε για κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχουμε το δικαίωμα να συζητούμε στο πλαίσιο αυτής της ε, συνέλευσης, χωρίς ίσως να έχουμε και τίποτα να λέμε, αλλά και η απλή ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών, οι που μπορούμε να απευθύνουμε στους συναδέλφους μας από τις χώρες ΑΚΕ, νομίζω ότι μπορούν παρόλα αυτά ε, να τους κάνουν τους ομολόγους μας να κινήσουν κάπως ε, τα πράγματα, να ταράξουν τα νερά στην κοινωνία ε, των πολιτών. Και νομίζω ότι και αυτοί ενθαρρύνονται και ενθαρρύνονται και από μια διάταξη της Συμφωνίας του Κοτονού που είναι η μόνη διεθνή συμφωνία, ήρθε στον παρόδο, η οποία με τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών ε, είναι υπέρ της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Δεν το συζητάμε παρελάχιστα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. Um, thank um, Σας ευχαριστώ. Μας υπενθύμισατε τις αδυναμίες και του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ε, χώρες εταίρους, αλλά, αλλά και το γεγονός ότι μέσω τη κοινή ε, κοινοβουλευτική συνέλευσης έχουμε μπορέσει να έχουμε απευθείας επικοινωνία, να βλέπουμε τι έχει γίνει στην πραγματικότητα και να ενημερωνόμαστε. Πράγμα το οποίο δεν ήταν δυνατόν στο παρελθόν να βλέπουμε δηλαδή που πήγανε τα χρήματα του EDF παραδείγματο του ε, Ταμείου Ανάπτυξη. Υπάρχουν ω εκ τούτου ζητήματα περίπλοκα. Είχαμε την ε, την κοινοβουλευτική συνέλευση των Ηνωμένες ε, τα ΕΠΑ, τι οικονομικέ ε, συμφωνίε σχέσης. Η Χίλερη Κλίντον εξέφρασε την προηγούμενη εβδομάδα αντιρρήσει για την συμφωνία για τον ειρηνικό. Είναι πολύ πιο περίπλοκα δηλαδή τα ζητήματα και την προηγούμενη εβδομάδα που συνομιλούσα με έναν πρέσβη από τις ε, χώρες του Ειρηνικού, από χώρα του Ειρηνικού, ε, με έβαλε στις σκέψεις για το Κοτονού, γιατί μου μίλησε για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνέπειες σε σχέση με τα τεκτενόμενα στα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη συμφωνία, γιατί τα κράτη της Συμφωνίας Κοτονού είναι και μέλη της ομάδας των 77 που δραστηριοποιείται σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Άρα αναπτύσσεται ένας ε, κόσμος διαφορετικός, όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Πολλές φορές θεωρούμε ότι την ε, σχέση αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιδιώκει ΑΚΕ, την επιδιώκουν τα κράτη ΑΚΕ. Μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, γιατί πριν από 30 χρόνια ίσως να μην είχαν άλλες επιλογές, ενώ τώρα έχουν νέους εταίρους. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη και αυτό, ότι υπάρχουν ε, επιλογές εταίρων διαφορετικών και εταιρικών σχέσεων. Ίσως να προτιμήσουν φερειπίν σχέση με την Κίνα. Κάποιες από τις χώρες αυτές που μπορεί να δώσει περισσότερα χρήματα κτλ. Στο παρελθόν κοιτούσαμε μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής βοήθειας και τώρα πρέπει να κοιτάξουμε με διαφορετικά μάτια την κατάσταση καθώς ο κόσμος αλλάζει, αναδύονται νέες ε, δυνάμεις. Είμαστε στην αρχή μια διαδικασία. Δεν ξέρω εσεί τι έχετε να προσθέσετε σε αυτό. Και βέβαια έχουμε και την Σεσίλ Κέγγε, συνάδελφο από την Μεκτή Επιτροπή, η οποία δυστυχώ όμω χρειάστηκε να φύγει, αλλά και άλλοι συνάδελφοι είναι εδώ που ίσω έχουν κάτι να προσθέσουν. Ο Λουί Μισελ Φερρυπίν δεν ήταν σε θέση να έρθει σήμερα, αλλά ξέρουμε ότι τον απασχολεί πολύ το θέμα αυτό και τον ε, παρακολουθούμε στην υπόθεση αυτή, ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσφορη έναρξη της περίοδου ε, μελέτης του τι θα γίνει μετά τη συμφωνία της Κοτονού στην επόμενη φάση. Καλωσορίζω τις πρώτες σας ε, συνεισφορές σε αυτά τα πρώτα στάδια μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς και ακόμη και αυτός ο σημερινός διάλογος είναι σημαντικός. Είναι μια σημαντική συνεισφορά στις δημόσιες διαβουλεύσεις. Εγώ έτσι το βλέπω. Είναι νωρίς για να δώσουμε διεξοδικές απαντήσεις στα ερωτήματα ή στα σχόλια που μόλις κάνατε. Όμως θα περιοριστώ στο εξή. θα επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα από τα πρώτα στάδια και ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες στη διάρκεια των διαβουλεύσεων στη συνέχεια. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των συμφωνίων Κοτονού ως τώρα. Οι πρώτες μου σκέψεις είναι ότι η Κοτονού ήταν αρκετά αποτελεσματική σε διμερές επίπεδο με τις επιμέρους χώρες δηλαδή και στις σχέσεις μας με αυτές αλλά ήταν ικανοποιητική και σε περιφερειακό επίπεδο. με οικονομικές κοινότητες, με κοινότητες δηλαδή χωρών που συνδέονται οικονομικά. Μα επέτρεψε λοιπόν να έχουμε και έναν δομημένο διάλογο με την Αφρικανική Ένωση, τη μεγαλύτερη από του περιφερειακού οργανισμού. Όμω, επίπεδο και ω ομάδα χωρών, τι βλέπω πιο πολλά μπορούσαν να έχουν κάνει για να αξιοποιήσουν το δυναμικό αυτή τη ομάδα χωρών, χωρών και. Βεβαίω. έχω κατά νου ότι η δέσμευση της ομάδας των χωρών και σε κάποια από τα διεθνή ζητήματα και σε κάποιες από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, λόγω χάρη για την νέα σειρά στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν η αφοσίωση των χωρών και ως ομάδας ήταν αρκετά περιορισμένη. Για το μέλλον λοιπόν, για την συμφωνία Κοτονού 2 ή όποια μορφή και αν πάρει αυτή, πρέπει ο συνολικός ρόλος της ομάδας των χωρών και να ενισχυθεί σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο. Και ο πολιτικός διάλογος και ο οικονομικός και ο εμπορικός πρέπει να ε, εντατικοποιηθεί. Και με τις χώρες της Αφρικής και της Καραϊδικής και του Ειρηνικού. Χρειάζεται λοιπόν μια σφαιρική δεσμευτική συμφωνία. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να βρούμε μια νέα αποτελεσματικότητα για τη Συμφωνία Κοτονού και να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες πιθανότητες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον και τα διαφορετικά πλαίσια σχέσεων που μπορεί να διαμορφωθούν. Η σαφέστερη ένδειξη που έχω εγώ ε, η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε από πολιτικής άποψης είναι ότι η επιστολή με την εντολή που μου ανέθεσε για τις θερμοδότητές μου ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούνκερ, στην αρχή της θητείας μου, εκεί λέγεται ότι στόχος μας, φιλοδοξία μας, είναι μια θεώρηση της συμφωνίας όχι τη συμφωνία με κεφαλαίο σίγμα, με μικρό. Να έχουμε λοιπόν διαπραγμάτευση για μια νέα συμφωνία ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτό είναι το σαφές για μένα. Είναι σαφής η πολιτική κατεύθυνση. Ακόμη και αν είναι κάπως ευρύ το πεδίο του εγγράφου σε σχέση με το όσο προβλέπει η εντολή, Ο στόχο είναι να συλλέξουμε στο δυνατόν περισσότερες απόψεις, ε, να τις συνθέσουμε και να μην περιορίσουμε αυτή τη στιγμή την ε, θεώρησή μας για το μέλλον προς μία και μόνη κατεύθυνση μπορεί, μπορεί να αφήσουμε την συμφωνία Κοτονού να εκπνεύσει χωρίς ε, να έχουμε προβλέψει το επόμενο στάδιο, για μένα αυτό αποκλείεται. Δεν είναι μια πιθανότητα που μπορούμε να δεχτούμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις διαφορετικές υποθέσεις που μπορούν να προκύψουν, αλλά θα ήθελα να μην καταλήξουμε σε αυτήν την ε, ε, αρνητική προοπτική. μια νέα μορφή τη συμφωνία επικαιροποιημένο περιεχόμενο ίσω είναι ένα νέο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ή να έχουμε μια πολιτική ομπρέλα. Μια πανοπλία μέτρων δεσμευτική και νομικός και με συγκεκριμένους γεωγραφικούς πυλώνες. Αυτό θα ήταν μια άλλη επιλογή, σαφώς, και ελπίζω αυτό να προκύψει από τις δημόσιες διαβουλεύσεις ε, και στην υπογραφή ε, συμφωνιών με τις υπόλοιπες χώρες και ε, στο ποράκι και τον Οι χώρες που δεν είναι μέλη της ομάδας ΑΚΕ ή την Κούβα. Η Κούβα είναι ΑΚΕ. αλλά δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κοτονού. Δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο νομικό πλαίσιο, όμως μπορούμε να τα επεξεργαστούμε αυτά μαζί. Θα προσπαθήσω επίσης να αναπτύξω τις απόψεις μου για κάποια από τα ζητήματα που εφήγησαν σήμερα στην πρώτη φάση των διαβουλεύσεών μας για την ένταξη στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να το προτείνει αυτό για, το επόμενο, για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2021 και μετά αλλά Υπάρχουν φυσικά πλεονεκτήματα και μενεκτήματα που θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να δούμε ποιο θα είναι ο πραγματικός αντίκτυπος τη ένταξη στον προπολογισμό του ΕΤΑ. Σε ό,τι αφορά την στάση της Επιτροπής, θα ακολουθήσουμε τα όσα έχουμε ε, αναλάβει για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με το ΕΤΑ. Θέλω όμως το μεταξύ να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη διαδικασία διαβουλεύσεων για την περίοδο μετά τη Συμφωνία της Κοτονού, προκειμένου να σκεφτούμε ποια θα είναι τα ωφέλη και το κόστο μια τέτοια διαδικασία. Βλέπω τώρα ότι η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια, η απλούστευση της δράσης μας, η περισσότερη, η μεγαλύτερη συνοχή της ε, αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διαδικασίας, η πολλή υλοποίηση, ο δημοκρατικός έλεγχος από την πλευρά του Προκοινοβουλίου, όλα αυτά είναι στοιχεία που υποστηρίζουν την ένταξη του ετάστον προπολογισμού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να φροντίσουμε και να δούμε ποιο θα είναι ο οικονομικό αντίκτυπο αυτή τη ένταξη στον προπολογισμό που σωστά μα υπέδειξε ο κ. Γκέρεντ. Θα ήθελα κάποια συζήτηση να γίνει για να αναδιαμορφώσουμε τη χρηματοδότηση των σχέσεών μας με τις χώρες ΑΚΕ και με μια νέα διάρθρωση, με νέα κριτήρια, ώστε τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν με διαφορετικό τόπο στον προπολογισμό. Θα χρειαστεί αυτό αφού θα συνεισφέρουν απευθεία στον προπολογισμό και όχι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο το ΕΤΑ να συμπιεστεί και να υπάρξει ένας ένα, να υπάρξει ένα κοινό χαρτοφυλάκιο, ένα κοινό ποσό που να είναι χαμηλότερο από το σημερινό ΕΤΑ. Επίσης μην ε, ξεχνάμε ότι και οι εταίροι μας των χωρών και έχουν αρνητική πρόσληψη ή μπορεί να εκλάβουν αρνητικά την ένταξη στον προπολογισμό αυτή ως υποβάθμιση των σχέσεών μας. Ε, ε, Συγκεκριμένες λοιπόν λύσεις μπορούν να συζητηθούν και να εξευρεθούν προκειμένου να υποστηρίξουμε τη συνολική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παραμείνει μια υψηλή προτεραιότητα στις αναπτυξιακούς μας στόχους η συμφωνία και για τις εμπορικές σχέσεις. Όχι, πρώτα απ' όλα για την πολιτική συνοχή και την ανάπτυξη. Το θεματολόγιο του 2030 με τους νέους ε, αναπτυξιακούς στόχους ε, εξυπακούει ότι θα πρέπει να υπάρχει σε μια σειρά από οριζόντια διασταυρούμενα θέματα ε, πολιτική συνοχή. Πρέπει να την εξασφαλίσουμε αυτή για την ανάπτυξη σε πολλά επίπεδα. Στις εσωτερικές μας πολιτικές δηλαδή τη δυνατότητά μας να εκπληρώσουμε τους ε, στόχους ανάπτυξης ε, διεθνώς. Πολιτική συνοχή λοιπόν στην εξωτερική μας δράση και αυτό είναι σημαντικό μέρος της συμβολής μας στην υλοποίηση των στόχων πέσιμης ανάπτυξης αλλά και συνοχή στην εσωτερική και εξωτερική διάσταση των σχέσεών μα. Οι εμπορικέ σχέσει είναι σημαντικέ για την πολιτική συνοχή. Είναι σημαντικό μέρο τη πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη. Απλώ θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Εάν μόνο οι εμπορικέ σχέσει ή οι διαπραγματεύσει, οι δασμολογικέ, οι συζητήσει περί κατάργηση δασμών ή μη δασμολογικών φραγμών είναι το υπέρτατος ε, στόχος των στόχων μας για την πολιτική συνοχή αρκεί να έχουμε νέα προτιμησιακά καθεστώτα για τους εταίρους μας των χωρών ΑΚΕ. Ή μήπως να δώσουμε ευρύτερο οικονομικό νόημα στις εμπορικές μας συμφωνίες. Με παρόμοια ή διαφορετικά εργαλεία. Πραγματικής οικονομικής σχέσης. Διότι οι εμπορικές σχέσεις έχουν βελτιώσει ή έστω απελευθερώσει μόνον, μάλλον δεν έχουν συμβάλει στο γεγονός, δεν έχουν συμβάλει στο να έχουν εμπορικά αγαθά, εμπορεύματα και υπηρεσίες να ανταλλάξουν οι εταίροι μας, που αυτό χρειάζονται πρώτα απ' όλα. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Οικονομικές σχέσεις που να βελτιώσουν τις βιομηχανικές τους δυνατότητες, τις δυνατότητες κατασκευής, το εμπόριο σε δίκαιους όρους, ε, Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, οι τελωνιακή δασμοί αλλά και η αποδυνάμωση των φυσικών του πόρων λόγω των εμπορικών διευθετήσεων είναι κάτι που θα το δούμε στο πλαίσιο των διεθνών πρωτοβουλειών για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των φορολογικών συστημάτων συνολικά το θεματολόγιο του 2020 συνέβαλε προς αυτό το σκοπό. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέραμε σε αυτό το σκοπό. Κάποιοι θα ισχυριστούν ίσως ότι δεν είμαστε έτοιμοι να προβλέψουμε και μια διεθνή εφορία όμως ως τώρα η συμβολή μας έχει βελτιώσει και θα συνεχίσει να βελτιώνει το πεδίο, τη συμμετοχικότητα, την ουσία και το περιεχόμενο της καλύτερης συλλογής φόρων διεθνώς. Συμβάλαμε σε αυτό το στόχο με την συνεισφορά μας τις ε, προτεραιότητες της Αντισαμπέμπα και της Νέας Υόρκης, με την ε, Φορολογική Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, με το εσωτερικό φορολογικό σύστημα που προβλέψαμε που είναι διαφανέστερο και με δεσμεύσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει. Contribute to, to, tax uh, avoidance, to, to, Η φοροαποφυγή θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την διάβρωση της φορολογικής βάσης και τις εκροές των, ε, των χρηματοπιστωτικών ε, εσόδων. Να πω και λίγα λόγια για τις σχέσεις μας με τις υπερπόντες περιφέρειες και διαμερίσματα. Ναι, ένα ειδικό δημοσιονομικό εργαλείο για αυτούς τους προορισμούς μας έχει απασχολήσει. Ήδη συζητήθηκε τη διαδικασία και τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όταν συζητήσαμε αυτήν την επταετία που διατρέχουμε, ήδη μας έχει απασχολήσει. Όμως, πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει σημαντικό. Πρέπει να εξεταστεί εν ώψη της διευθέτησης και του πλαισίου για μετά το 2020. Η Επιτροπή είναι έτοιμη. Θέλει να υπάρξει επικοδομητικός διάλογος για ένα ειδικό δημοσιονομικό εργαλείο για τις περιπόντες περιφέρειες και διαμερίσματα. Έχουμε περίπου 65 εκατομμύρια για αυτές τις περιοχές και 11 μόνο από το ΕΤΑ, αν και είναι σημαντική αύξηση για το ΕΤΑ. Να πω αυτό το χαρτοφυλάκιο πρόκειται να διαφυλαχθεί και ως προς το ύψος του. Και ως προς τις πολιτικές μας δεσμεύσεις για να στηρίξουμε τις στρατηγικές και τις πολιτικές των υπερπόντιων περιφερειών και διαμερισμάτων. Βεβαίω η συζήτηση αυτή μπορεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το 11ο ΕΤΑ. Γιατί έχει κλείσει αυτή τη στιγμή η συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο και τη δικασία έχει ξεκινήσει. και σε δημερές και σε περιφερειακό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προγραμματισμού εντός του 2016 θα έχουμε και διεξοδικές διαβουλεύσεις για το πώς να προχωρήσουμε σε ένα ειδικό ε, χρηματοδοτικό εργαλείο για τις περπόντες περιφέρειες και διαμερίσματα. Καλωσορίζω λοιπόν τη δέσμευση και την αφοσίωση των μελών της Επιτροπής ΔΕΒΕ στην όλη διαδικασία για την αναδιαμόρφωση του πλαισίου μετά την πρώτη φάση της Συμφωνίας Κοτονού. Μιλήσαμε για τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Είδαμε ποιες είναι οι καταστάσεις που μπορεί να διαμορφωθούν θα φροντίσουμε όταν πάρουν σαφέστερη μορφή να ε, εξορθολογήσουμε τις προτάσεις μας και ανάλογα με το τι θα προκύψει από τη διοικασία διαβουλεύσεων με τις χώρες ΑΚΕ. Αναμένουμε οι εταίροι μας από τις χώρες ΑΚΕ να εκφράσουν και αυτοί τις δικές τους ε, προτεραιότητες θα υπάρξει και ομάδα εργασίας που ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα και ελπίζω ότι ως το τέλος του 2016 θα έχουμε πλέον και την ανακοίνωση στα χέρια μας. Ακόμη και αν η μελέτη αντικτύπου ακολουθήσει και συμβαδίσει όλη αυτή την προσπάθεια, με αυτή την προσπάθεια. Αρχές 2017 πάντως μάλλον θα φτάσουμε στο επίπεδο της ανακοίνωσης και θα αποφασίσουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να είμαστε καλώς προετοιμασμένοι για την φάση και τις διαπραγματεύσεις μας μετά την Κοτονού. Okay. Okay. Σας ευχαριστούμε. Και τελειώσαμε ακριβώς στις 5 η ώρα. Μας δώσετε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να παρακολουθήσουμε, να συζητήσουμε. Γιατί προσέτα τα συμπεράσματα ήταν πολύ καλή αρχή η σημερινή και σε ευχαριστούμε θερμά. Συνάδελφοι, η προσοχή μας συνεδρίες προβλέπεται για τι 9 Νοεμβρίου 3 το απόγευμα, 10, 10 Νοεμβρίου πρωί και απόγευμα. Θα τα πούμε βέβαια το μεταξύ και στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ.